May I ask you, colleagues, to take seat? I will give a couple of minutes uh, during. Λοιπόν, θα δώσουμε λίγα λεπτά στην υποψηφία επίτροπο αλλά και στους δημοσιογράφους για να πάρουν τις φωτογραφίες και μετά θα τους ζητήσω να φύγουν από την αίθουσα ή μάλλον να καθίσουν κάπου αλλού. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν. Να σας καλωσορίσω κυρία Βέσταγκερ εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Είναι η τρίτη ακρόαση που διοργανώνει η Επίτροπη ΕΚΟΝ. Έχουμε γίνει μηχανή ακροάσεων, αλλά είναι μεγάλη σημασίας. Προσπαθούμε να αξιολογήσουμε λοιπόν τους προτινομένους επιτρόπους και στο σύνολό τους και μεμονωμένα επί τη βάση των αρμοδιοτήτων τους, της ευρωπαϊκής τους αφοσίωσης και της ανεξαρτησίας τους της προσωπικής από διάφορα συμφέροντα και φυσικά να αξιολογήσουμε και τις πολιτικές τους προτεραιότητες και τη δυνατότητα συνεισφοράς τους στο νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι κανόνες μας είναι οι εξής. Η υποψηφία επίτροπος θα κληθεί να κάνει μια εισαγωγική παρουσίαση 15 λεπτών το πολύ. Και αμέσως μετά θα υπάρξουν 45 ερωτήσεις, ένα λεπτό για την ερώτηση και δύο λεπτά για την απάντηση. και στο τέλος θα υπάρξουν ε, ομιλίες από τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων. Θα ζητήσω από όλους τους ομιλητές παρακαλώ να σεβαστούν το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Ένα λεπτό και μετά δύο λεπτά όπως είπα η απάντηση. Η διευμηνία παρέχεται σε 23 γλώσσες. Αλλά θα ήθελα να ζητήσω και από τους ομιλητές παρακαλώ να μην ομιλείτε πάρα πολύ γρήγορα και να σας διαβεβαιώσω ότι η συζήτηση αυτή θα μεταδοθεί από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν δώσω το λόγο λοιπόν στην υποψηφία επίτροπο, να πω ότι εμείς ε, προωθούμε σαν στόχο την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίω. Είναι ένας ιστορικός στόχος αν θέλετε και έχει πολλές αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα αυτό αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε τις δυνατότητες αυτές και στο, στο βαθμό του εφικτού βέβαια κάθε φορά να μπορέσουμε να παίρνουμε αποφάσεις με βάση τη σωστή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η λειτουργική μορφή του ανταγωνισμού σε τομείς όπως τα χρηματοπιστωτικά και οι νέες τεχνολογίες θα συνεισφέρει τα μάλα στην ανάπτυξη και στην απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη και τον ανταγωνισμό από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε όπως το θέμα των κρατικών μονοπωλίων, τα προβλήματα του πιστοτικού τομέα ε, και ο ενιαίος μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Λοιπόν, θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία ε, Μαγκρέτε Βέισταγκερ για την παρουσίασή της.